Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω και μια αντιπροσωπεία της Καναδικής Βουλής. Προεδρεύεται η αντιπροσωπεία του Καναδά Προεδρεύεται λοιπόν έλεγα από από τον πρόεδρο της ε, διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας Ευρώπης Καναδά και περιλαμβάνονται βουλευτές ε, και ε, γερουσιαστές από, όλες, όλα τα κρατήδια του Καναδά, από όλες τις πολιτείες καλύτερα του Καναδά. Βρίσκονται εδώ με αφορμή την 30 συνάντηση την διακοινοβουλευτική ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά. Εμείς εκφράζουμε και τη λύπη μας για τα τριγικά γεγονότα στις 2 Οκτωβρίου γύρω από την Βουλή στην Οτάβα. Εκφράζουμε ε, την αλληλεγγύη μας και το θαυμασμό μας για τον οποίο, με τον οποίο ε, για το φάρος μάλλον και την αξιοπρέπεια με την οποία αντέδρασαν οι Καναδοί επί τη βάση των κοινών αξιών που πιστεύουμε στον Καναδά και στην Ευρώπη. Έχουμε ε, μακρότερες σχέσεις ανάμεσα στο δικό μας κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο της Οτάβα και τους καλωσορίζω αγγλικά και γαλλικά για μια ακόμη φορά. Περνάμε πλέον στις ψηφοφορίες. Η Αγιάλα Σεντέρ έχει το λόγο. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Δεν ξέρω εάν αυτό ε, σήμερα το πρωί ε, το είπατε. Ε, θα πρέπει όλοι να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την πρόσδεση στο κομίτη της Ροσέτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει να το καλωσορίσουμε και να το χαιρετήσουμε. Ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα της ευρωπαϊκής τεχνολογίας και βιομηχανίας και συμμερίζομαι αυτό που είπατε κυρία Γιάλα Σέντερ. Και το λέω αυτό και σαν τέος επίτροπος υπεύθυνο για τη διαστημική πολιτική. Περνάμε στην έκθεση Χάουταλα. Πρόταση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Υπέρ